Chers collègues, je vous propose que nous euh, Να ξεκινήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν υπάρχουν ε, σχόλια, φαντάζομαι, πάνω στη μερίσια διάταξη. Και αφού δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, υιοθετείτε. Δεν έχω ανακοινώσεις ε, της Προέδρου. Πάμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, εξέταση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων αφορά την αναθεώρηση της διαδικασίας για την μόνιμη αυτή διαρθωμένη συνεργασία. Καλώς ήρθαν οι προσκεκλημένοι μας. Ο κύριος Αγνού Μολενάρ, ε, επικεφαλής του ΣΕΚΤΕΛΦΟΠ, ο κύριος Αλεξανδρινός Σινιώνη, ε, τμήματάρχης του ΣΕΣΠΕ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Άμυνας, και ο κύριος Μολνή, διευθυντής, ε, υποδιευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και Στατηγικών Σχέσεων. Η, η συνεργασία αυτή υπάρχει στην συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, για μια, ένα πυρήνα των κρατών να αναπτύξουν περισσότερο την ε, άμυνά τους. Ε, προβλεπόταν να ξεκινήσει το 2010 και τελικά ενεργοποιήθηκε το 2017 για 25 κράτη-μέλη. Ε, είναι προωθεί την ε, πολιτική ασφάλειας και κοινή άμυνας και βασίζεται στην διαφοροποιημένη ε, ένταξη. Ε, αφορά όλα τα κράτη-μέλη και η μόνη δεσμευμένη συνεργασία επιτρέπει σε μια ομάδα χωρών, όταν το επιθυμούν, να έχουν πιο δεσμευτικές μια πιο δεσμευτική στάση σε ό,τι αφορά την άμυνα και να συμμετέχουν στα προγράμματα εξοπλισμού συνεργα... σε... στα πλαίσια μια ευρωπαϊκής συνεργασίας, ενισχύοντας ε, την επιχειρησιακή δράση των στρατών τους. Ε, κοινοποιήθηκε το 2017 ε, με 20 δεσμεύσει, δεσμευτικές. Ε, έχουμε το Δεκέμβριο του 2017 παρουσιάστηκαν ε, τα πρώτα, ένα μια πρώτη λίστα ε, σχεδίων, project, ε, για κράτη άλλη μέλη και εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2018. Ένας οδικός χάρτης που αφορά τη λειτουργία του, της διαστομένης συνεργασίας υιοθετήθηκε το Μάρτιο του 2018. Εν συνεχεία 17 νέα project υιοθετήθηκαν τον Νοέμβριο του 2018 και άλλα 13 το, στις 12 Νοεμβρίου του 2019 και τελικά έχουμε 47 ουσιαστικά τέτοια σχέδια για την μόνιμη διαφθομένη συνεργασία. Η ύπατη εκπρόσωπο τη ε, Ένωση για την Εξωτερική Πολιτική και Άμυνας παρουσίασε τον Μάιο του 2019 την πρώτη έκθεσή τη για την εφαρμογή τη μόνιμης διεθνωμένης συνεργασία ε, και το Συμβούλιο υιοθέτησε στι 6 Μαου του 2016 τις συστάσεις αυτέ, λαμβάνοντα υπόψη τι προτάσει στην έκθεση. Ε, είμαστε σε μια φάση λοιπόν τώρα όπου πρέπει να αξιολογήσουμε την διαθωμένη συνεργασία, να δούμε τι, δυνατά στοιχεία έχει, τι αδυναμίε έχει και να δούμε πού πώς θα προωθηθεί στο μέλλον. Η επιτυχία της βασίζεται στις ε, συνεισφορές των κρατών και τους επιτρέπει να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους ε, πιο, πιο δεσμευτικό τρόπο στους πέντε τομείς ε, που, βασίζουν, που καθορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλου 10 ε, που θεσπίζει την ε, μόνη διεθνή συνεργασία. Ο σεβασμό αυτών των ε, δεσμεύσεων μα επιτρέπει να αυξήσουμε τι δυνατότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στρατηγική τη αυτονομία. Πρέπει να διαρωτηθούμε. Αυτοί οι στόχοι έχουν υλοποιηθεί, ποιοι είναι, είμαστε στο δρόμο. Τα κράτη-μέλη σέβονται τα, τους όρους για τις δαπάνε σε επίπεδο επενδύσεων, σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό τη άμυνα, ε, συντονίζουν τις πολιστικέ άμυνά τους και εναρμονίζουν τις ε, ανάγκες τους. Και επίσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον εξοπλισμό από κοινού, ε, σε ό,τι αφορά την κατάρτιση ας πούμε, του προσωπικού, το, την επιμελητία κτλ. Ε, επίσης, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος τέλη Μαρτίου του 2020 θα παρουσιάσει τη δεύτερη έκθεση για τη μόνιμη διεθνή συνεργασία και θα, αυτό θα είναι ε, το σημείο φετηρίας ε, για τη στρατηγική αναθεώρηση για να ετοιμάσουμε τον απολογισμό ε, για την περίοδο 2021-2025. Το Συμβούλιο θα υιοθετήσει συστάσεις προς τα κράτη-μέλη το Μάιο του 2020. Στην τελευταία φάση, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ε, και Άμυνας, ε, τέλη φθινοπόρου, ε, θα γίνει μια διαδικασία αναθεώρησης απόφασης του Συμβουλίου του 2017 που καθόριζε τη δεύτερη σειρά στόχων για την περιοδο 2021 2021-2025. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ετοιμάσει μία σύσταση. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Ραντοσλάβ Σικόφσκι του ΕΛΚ. Γι' αυτό ακριβώς συνεδριάσουμε σήμερα για το θέμα αυτό. Ξεκινώντα λοιπόν, θα ήθελα ο κύριο Μολενάρ να πάρει το λόγο, ούτω ώστε να μα παρουσιάσει τη διαδικασία στρατηγική αναθεώρηση τη μόνιμη διαθμένη συνεργασία, τη μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για να κάνουμε αυτή την αναθεώρηση και τα πρώτα συμπεράσματα στα οποία φτάσατε. Θα δώσω ε, συνεχεία το λόγο στον λοχαγό Σούμαν ε, από την ε, του Αρχηγείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μας μιλήσει για τους τελικούς χρήστες που είναι οι στρατιωτικοί ε, και συνεχεία ε, στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Άμυνα μέλο τη γραμματεία του, της Μόνιμης συνεργασία και στον κύριο Μουλνή για να μα εξηγήσει πώ η Μόνιμη Θερμανική Συνεργασία συνδυάζεται με άλλε ευρωπαϊκέ πρωτοβουλίε και πώ μπορεί να καθορίσει περισσότερο την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Ο κύριος Μολενάρ θα μιλήσει καταρχάς για 5 με 7 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνεται να σας ενημερώσω για το πώς έχει κατάσταση με τη στατική αναθεώρηση της μόνιμης διαδρομένης συνεργασία, που είναι ορόσημο για τη φετινή μας δουλειά. Και σημαντικό βέβαια είναι να τηρήσετε ενήμερη ω Κοινοβούλιο για τι εξελίξει στο πλαίσιο αυτή τη διαδικασία και προσβλέπω και στην ανταλλαγή απόψεων που θα ακολουθήσει. Όπω ξέρετε, συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο τη γραμματεία ε, τη ΠΕΣΚΟ, η ΕΔ, ε, για την ασφάλεια και την άμυνα του συγκεκριμένου τμήμα από τη δική μα πλευρά. Σίγουρα 25 συμμετέχουσες χώρες ε, είναι αυτές που έχουν τα αρμοδιότητα. Η νομική βάση για τη σαπτική αυτή αναθεώρηση ήταν η απόφαση ίδρυσης με στόχο τη βελτίωση, η αναθεώρηση πιο δεσμευτικών ε, δεσμε... υποχρεώσεων. Και εσείς αναφερθήκατε στις διάφορες προθεσμίες. Η πρώτη φάση λίγη φέτος, έχουμε την άλλη από το 2021 στο 2025, και έπειτα θα οριστούν πιο ακριβώ τα επόμενα στάδια. Θα πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη η πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των δεσμεύσεων τη ΠΕΣΚΟ και το μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλεία. Ε, θα έλεγα ότι συνολικά πρέπει να ξέρουμε ότι το Δεκέμβριο του 2017, όπως αναφέρεται, δηλαδή σύντομα, ε, πρόσφατα ε, θεσπίστηκε αυτή η συνεργασία. Χρειάζεται αναθεώρηση, θα πρέπει όμως ε, χωρίς να πάμε σε μια άρθρη αναθεώρηση να δούμε πού μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα για να προχωρήσουμε. Και βέβαια προτεραιότητα, ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, θα ήθελα να σας πω ευθύ εξ αρχής ότι σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τρίτων κρατών, υπό ποιες προϋποθέσεις ε, τρίτα κράτα μπορούσαν να κληθούν να συμμετέχουν σε project, Τη ΠΕΣΚΟ είναι κάτι το οποίο κρεμεί ακόμη. Η εκπεριτροπή στην Προεδρία αυτή τη στιγμή η Κροατία είναι αυτή η οποία καλείται να βρει λύσει. Ε, πέρυσι σημειώθηκε πρόοδο, χωρί όμω να έχει ακόμη υπάρξει συνένεση. Δεν εντάσσεται το θέμα όμω στην φετινή στρατηγική αναθεώρηση. Είναι ένα άλλο σάξονα, σημαντικό και αυτό, βέβαια. Και τι επόμενες εβδομάδε νομίζουμε θα έχουμε κάποιε εξελίξει. Υπάρχει διαθρωμένη διαδικασία στο πλαίσιο της γραμματείας, της ΠΕΣΚΟ μαζί με τα κράτη-μέλη με στόχο να δούμε τι βελτιώσεις ε, μπορούμε να επιφέρουμε γιατί αυτή τη στιγμή είναι, ε, ακόμη είμαστε στην πρώτη φάση, λέγουμε τις ιδέες των κρατών μελών. Το δεύτερο βήμα, το δεύτερο στάδιο, θα είναι από τον είπα εκπρόσωπο πλέον να, έχουμε συστάσεις ε, στην ετήσια έκθεση για, το, για την κατάσταση εφαρμογής της ΠΕΣΚΟ. Μάρτιο, αρχές Απρίλιο θα του λάβει το Συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια θα δώσει καθοδήγηση στο πλαίσιο των συμπερασμάτων και των συστάσεων που θα πρέπει να εγκριθούν το Μάιο γιατί την μόνιμη να είναι Το επόμενο βήμα θα επανεξεταστούν οι πράξει πράξεις για να αντικατοτρίζονται οι αλλαγέ και οι νέε συμφωνίε μέχρι τα τέλη του έτου. Με τη θέση πια παράδειγμα, ε, μάλλον με αυτή τη συμφωνία ίδρυση, να δούμε αν υπάρχουν ε, αλλαγέ. αν χρειάζεται μια νομική τροποποίηση και έχουμε και την απόφαση του Συμβουλίου για τους κοινού κανόνες διακυβέρνησης ε, των σχεδίων. Και έχουμε φτάσει ήδη στο επόμενο έτος. Οπότε και θα δούμε συγκεκριμένα τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί και οι οποίοι θα καθοδηγούν τα σχέδια εφαρμογή για τις διάφορες δεσμεύσεις. Ένα ακόμη βήμα της διαδικασίας. Μετά την αναθεώρηση της μόνιμης διθρωμής συνεργασίας, αλλά σημαντικό και αυτό. για τον πιο απακριβή ορισμό των ε, δεσμεύσεων για την επόμενη φάση της ΠΕΣΚΟ. Σε αυτή τη διαδικασία, μαζί με τα κράτη-μέλη, εξετάζουμε τρει τομεί, τι δεσμεύσει, ε, τα έργα, οι σχέδια και τις διαδικασίε. Είπατε και εσείς σωστά, κυρία Πρόεδρε, ότι στόχος μας είναι να ανοίξει δρόμο για την επόμενη φάση της ΠΕΣΚΟ. Και ένα πολιτικά πολύ ευαίσθητο σημείο εδώ είναι να ε, βρεθεί ποιο είναι το απτό παραδοτέο αποτέλεσμα που θέλουμε για τα επόμενα χρόνια από πλευρά ΠΕΣΚΟ. Είναι σημαντικό για την εξοπιστία τη ε, μόνιμη διαθρωμένη εργασία. Έρχομαι στου διάφορου τομεί. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τι δεσμεύσει. Εδώ πρέπει να είμαστε κάπω ρεαλιστικοί, υπό την έννοια ότι τα κράτη-μέλη αρχίζουν ε, να ε, κάνουν κτήμα του σιγά-σιγά αυτές τις δεσμεύσει. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να μην μπρούμε σε δραστικέ αλλαγέ σε αυτό το σημείο. Δεύτερον, εστιάζουμε στο συντονισμό, στην εφαρμογή, στην υλοποίηση. Και έχουμε και την ετήσια έκθεση του προσώπη για την ΠΕΣΚΟ που επίκειται και που θα είναι ένα σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδικασία. Θα μετρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Τρίτο σημείο, και ήδη αυτό εντάσσεται και στη συζήτηση που γίνεται, είναι να εστιάσουμε περισσότερο Στι επιχειρησιακέ, του καλούμενε δεσμεύσει, για την ενίσχυση τιμότητα ε, τη συμβολή, ε, στι διάφορε επιχειρήσει τη ΚΕΠΑ. Πρέπει να γίνουν περισσότερα σε αυτό το πεδίο. Είναι προφανέ. Και αν δεν μπορούμε την επικαιροποίηση να την δούμε στι ε, δεσμεύσει, μπορούμε ίσω να χρησιμοποιήσουμε του πιο συγκεκριμένου αυτούς στόχου για να δώσουμε πιο αναλυτική καθοδήγηση. Ό,τι αφορά τα έργα σχέδια. Έχουμε 47 τον αριθμό και το βασικό είναι ότι πρέπει να παραμείνουμε εστιασμένοι, πρέπει να υπάρξει πρόοδο για την ανάπτυξη των αναγκαίων δυνατοτήτων και βελτίωση τη ετοιμότητα. Δεύτερον, και επειδή έχουμε και μεγάλο όγκο σχεδίων έργων, το θέμα πλέον είναι να μπορούμε να το ομαδοποιήσουμε, να έχουμε κλάστερ για να έχουμε περισσότερε συνέργειε. Παραδείγματο χάρη, αντικειτική μέρημνα, κινητικότητα ή κυβερνοχώρο ασφάλεια. Κάτι που αφορά κυρίως τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν. Θα σας τα πει και ο Αλεσάνδρου στη συνέχεια. Διαδικασίε και μέθοδο εργασία τρίτο τομέα. Το βασικό εδώ είναι πώ θα επιγραμμίσουμε τη διαδικασία τη ε, ΠΕΣΚΟ με, την, το λεγόμενο CARD, την ενιαία εξολόγηση που έχει το δικό τη ρυθμό και το δικό του ε, κύκλο λήψη αποφάσεων. Και έχουμε και το Ταμείο Άμυνα που εξαρτάται από τα σχετικά προγράμματα εργασία. Ένα άλλο θέμα για τι διαδικασίε και τη μέθοδο εργασία είναι πώ θα ενισχύσουμε την εκτίμηση και θα αυξήσουμε την προσθέμενη αξία και στι και για το μέλλον σε ό,τι την πρόοδο των διαφόρων έργων σχεδίων. Βεβαίω και εστιάζουμε στην πρόοδο τη ΠΕΣΚΟ, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το δούμε μεμονωμένα. Πρέπει να υπάρξει συνεκτικότητα με άλλε αμυντικέ πρωτοβουλίε, CARD, ε, ETF. Τα ανέφερα αυτά, είναι σημαντικά και λαμβάνονται υπόψη την αναθεώρηση της ΠΕΣΚΟ. Και, το HR... Ε, και ο υπάτος εκπρόσωπο, έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ω υπεύθυνο μαζί και με το Σώμα των Επιτρόπων εν γέννη. Πέραν όμω, των αμυντικών μέσων και εργαλείων, ίσω θα πρέπει να δούμε με ποιου άλλου τρόπου η ΠΕΣΚΟ προ... Ε, μια διασύνδεση με κάποιες άλλες αμυντικές πρωτοβουλίες που δεν υπήρχαν όταν ιδρύθηκε η ΠΕΣΚΟ, αλλά σιγά σιγά έχουν αναδυθεί, έχουμε το ευρωπαϊκό την μηχανισμό ασφάλειας, ε, τις στρατιωτικές δυνατότητες και την θαλάσσια ασφάλεια, τις ευρωτικές απειλές, κλίμα και άμυνα, πρόσφατη πρωτοβουλία. Ολοκληρώνοντας, ποιο είναι το βασικό μήνυμα. Πράγματι, τα κράτη-μέλη έχουν δημιουργήσει ένα μοναδικό εργαλείο βάσει τη συνθήκη για μια πιο δεσμευτική συνεργασία μεταξύ των 25 κρατών μελών. Είναι κάτι μοναδικό, δεν υπάρχει κάπου αλλού, παρά μόνο σε ενωσιακό επίπεδο. Είναι η ΠΕΣΚΟ λοιπόν ένα πολιτικό πλαίσιο στενότερη συνεργασία στον τομέα τη άμυνα. Εξού και το πρώτο και βασικότερο είναι να παραμείνει αυτό ο ρυθμός. Ε, υπάρχουν στρατιωτικοί, πολιτικοί στρατηγική, οικονομική και άλλοι λόγοι που είναι πάντα επίκαιροι. Και Σίγουρα, επειδή μόλις πριν δύο χρόνια δημιουργήθηκε αυτή η μόνιμη διαφωνή συνεργασία, πρέπει να του δοθεί παραπάνω χρόνος. Εμείς από την πλάτη της Γραμματείας θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη, ώστε να έχουμε αυτά αποτελέσματα και να συνεχίσουμε το δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Να κάνουμε πιο ισχυρή και πιο ασφαλή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον πλήρχο Λάρς Σούμαν από το ε, τμήμα του στρατιωτικού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και να σας ευχαριστήσω και για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας απευθύνω το λόγο σήμερα εδώ. Μετά από τον κύριο Μολενάρ και την ε, πλήρη εισαγωγή των όσων κάνουμε αυτή τη στιγμή στην ΠΕΣΚΟ και ο κύριος Τσιγκιόνι θα σας ενημερώσει ε, για τα προγράμματα. Εγώ θα επικεντρωθώ σε κάποιες στρατιωτικές πτυχές προφανώς. Αυτό το οποίο έχει σημασία εν τέλει είναι πώς ε, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το στρατιωτικό μέσο επιτυχώς όταν θα χρειάζεται. Πώς θα συντονίσουμε τις επιχειρήσεις μας, πώς θα πληρούμε τις απαραίτητες απαιτήσει και πώς ε, θα στελεχώσουμε ε, τα σώματό μας. Ε, Λαμβάνοντα υπόψη ε, την κατάσταση αυτή τη στιγμή, έχουμε ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωση. Επομένω, δεν πρόκειται για μια θεωρητική διαδικασία. Πρόκειται για κάτι συγκεκριμένο, το οποίο συζητούμε για την ασφάλεια των ανδρών και γυναικών που έχουμε στο εξωτερικό ανα πάσα στιγμή προκειμένου να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα, θα πρέπει να γίνει μια ολιστική συζήτηση, όπου θα θέλαμε εν τέλει να καταλήξουμε μέσω της ΠΕΣΚΟ. Να δούμε δηλαδή ποιος είναι ο τελικός στόχος της ε, ΠΕΣΚΟ. Είναι να μετρήσουμε πού βρισκόμαστε και να δούμε τι πρέπει να προσαρμόσουμε. Όχι μόνο για τη στρατηγική αναθεώρηση, αλλά τακτικά και στις αιτήσεις εκθέσεις ε, της ε, στρατηγικής αναθεώρησης. Αυτή τη στιγμή η στρατηγική αναθεώρηση είναι κατάλληλη για να δούμε αν γίνονται σωστά τα πάντα και την κατάλληλη στιγμή και αν είμαστε στο σωστό δρόμο. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε συνέργειες με άλλες αμυντικές πρωτοβουλίες και άλλες διαδικασίες. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι έχουμε επιτύχει ήδη μέχρι τώρα και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε τις προσπάθειές μας. Από στρατιωτική σκοπιά πρέπει να επικεντρωθούμε στην επίτευξη του ε, στρατιωτικού επίπεδου φιλοδοξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση της, του Συμβουλίου που καθορίζει την ΠΕΣΚΟ αναφέρεται σε ένα πλήρες πακέτο που θα πρέπει να είναι και ο τελικός μας στόχος. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να αρχίσουμε να καθορίζουμε τι εννοούμε ε, με αυτό. Και πιστεύω ότι το στρατηγικό σύμφωνο, που είναι μια πρωτοβουλία που συζητιέται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο, είναι ένας τρόπος να έχουμε και μια πιο ε, σαφή άποψη από αυτό. Βραχυπρόθεσμα αντιλαμβανόμαστε καλά ποιε είναι οι απαιτήσει μα σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο προγραμματισμού για να δούμε και τι ικανότητέ μα τι απαιτήσει χρειαζόμαστε και τους ε, βασικούς στόχους υψηλού αντικτύπου που είναι τα βασικά και να που έχουμε αυτή τη στιγμή και τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουμε και ως πηξίδα για να δούμε πού θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις ε, προσπάθειές μας. Αν τα καταφέρουμε εκεί, ίσως θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε ε, γενικότερα στα θέματα αυτά. Γι' αυτό και ακριβώς οι επιχειρησιακές απαιτήσει οι 12, 13 και 14 θα πρέπει να ενισχυθούν. Υπάρχουν νέες προτάσεις ε, σχεδίων, οι οποίες θα πρέπει να επικεντρωθούν όλο ένα και περισσότερο για το πώς μπορούμε να μειώσουμε τα κενά που έχουμε στις ικανότητές μας, προκειμένου να μπορέσουμε να μετριάσουμε και τα ε, ελαττώματά μας. Και έτσι η ΠΕΣΚΟ θα ε, επικεντρωθεί καλύτερα στα αποτελέσματα, όπως έχουν ζητήσει και πολλοί από τους συμμετέχοντες. Πρέπει να βελτιώσουμε τις διαδικασίες και αυτό ίσως θα μπορούσε να γίνει και με διασύνδεση υφιστάμενων δυνάμεων για να μπορέσουμε να τις έχουμε διαθέσιμες για τις παρούσες αποστολές και επιχειρήσεις μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 47 προγράμματα και ίσως θα πρέπει να τα ομαδοποιήσουμε και να έχουμε παρόμοια προγράμματα μαζί σεβόμενοι φυσικά και τις προϋποθέσεις που έχουν εκφράσει τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν και αυτή θα πρέπει είναι μια διαδικασία που θα ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω και κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να προχωράει αυτόνομα. Εμείς όμως ε, θα πρέπει να υποστηρίζουμε και αυτά τα, ε, τη διαδικασία. Και τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι η συμμετοχή της Στρατιωτικής Επιτροπής σε κάθε στάδιο τη διαδικασία στρατηγικής αναθεώρησης θα επιβεβαιώσει ότι η ΠΕΣΚΟ είναι μια πρωτοβουλία άμυνα τελικά η οποία θα ε, μπορέσει να επιτρέψει και την κατάλληλη χρήση στρατιωτικού επίπεδου φιλοδοξία και τη χρήση της στρατιωτική ικανότητας τη ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Αλεσάνδρο Τσινιόνι από, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την πρόσκλησή σας να μιλήσω για την μόνιμη διαρθωμένη συνεργασία στην, Επιτροπή, στην Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας, μαζί με τους συναδέλφους μου. Θα ήθελα να εστιάσω στις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τα σχέδια. Όπως θα ξέρετε, ε, το τελευταίο τμήμα σχεδίων ε, υιοθετήθηκε το Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2019 με 13 νέα project στα, που προσθέθηκαν στα υπάρχοντα 34. Τα 10 από τα 13 αφορούν την κατάρτιση και εκπαίδευση. Τα σχέδια ΠΕΣΚΟ θέλουν να δώσουν αποτελέσματα σημαντικά για τις ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να υπενθυμίσω πώς επιλέγονται αυτά τα σχέδια από τους, τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη στη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Το πρώτο βήμα είναι η υποβολή προτάσεων από τα κράτη-μέλη για σχέδια. Τα κράτη-μέλη ε, μιλούν με άλλα κράτη-μέλη για τα σχέδιά τους για να δημιουργήσουν μια κάποια συνένεση. Ε, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη και η πρόταση για σχέδιο υποβάλλεται στη γραμματεία προς αξιολόγηση, στην, γραμματεία της ΠΕΣΚΟ, ε, που την κάνουν οι συνάδελφοι ε, από επιχειρησιακή σκοπιά. Και η εκτέλεση γίνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας που ασχολείται με τα θέματα των ε, δυνατοτήτων. Εξετάζουν τη συνοχή, την οριμότητα του, σχεδίου, συνάφεια με τον ΝΑΤΟ και τα οικονομικά στοιχεία. Η οριμότητα του σχεδίου είναι σημαντική αφορά το αν υπάρχουν αρμονισμένες προϋποθέσεις που είναι σημαντικές για να ξεκινήσει μια συνεργατική προσπάθεια και αν υπάρχει ένας καλός οδικός χάρτης για την εναρμόνιση αυτών των project. Με βάση την αξιολόγηση που γίνεται βάση των προτάσεων από τη Γραμματεία της Μόνιμης Διαθρομένης Συνεργασίας, τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη θα επιλέξουν στο Συμβούλιο τα σχέδια τα οποία θα αναπτύξει η μόνιμη διαφωμένη συνεργασία. Πώς παρακολουθούμε τώρα ότι αυτά τα σχέδια προχωρούν όντως. Αυτό είναι βασικό θέμα, το οποίο εξετάζεται και στη στρατηγική αναθεώρηση της μόνιμης διαφθομένης συνεργασίας. Προς το παρόν, μια αυτοαξιολόγηση για την πρόοδο γίνεται από τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στα σχέδια αυτά. Τα κράτη-μέλη κάνουν λοιπόν αυτή την αξιολόγηση που συμμετέχουν στο project. Με βάση την απόφαση του Συμβουλίου για τις, ε, τους κανόνες διαχείρισης των project του ΠΕΣΚΟ, το Συμβούλιο ενημερώνεται από τα κάτι μελη που συμμετέχουν για τις εξελίξεις του συγκεκριμένου σχεδίου άπαξ ε, ετησίως. Αυτές οι εκθέσεις έχουν ε, παγιες, παγιοποιημένες πληροφορίες για την πρόοδο που έχει γίνει προς, με σκοπό την εφαρμογή του project, τον οδικό χάρτη, τους στόχους και τα ορόσημα και η συνεισφορά στην υλοποίηση των πιο σημαντικών δεσμεύσεων που αφορούν τη μόνιμη διαθεμένη συνεργασία. Οι νέε εκθέσεις θα σταλούν από εμά τη Γραμματεία στο Συμβούλιο στα τέλη του μήνα από ό,τι προβλέπουμε. Επίσης, θα είναι σημαντική η συνεισφορά για την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή των σχεδίων ΠΕΣΚΟ ε, που θα γίνει ε, τέλος Μαρτίου. Θα ήθελα τώρα να τονίσω κάποια σχέδια για να δείτε πόσο ποικίλα είναι σε ό,τι αφορά την κλίμακά τους, τη συμμετοχή τους, αλλά και τη φιλοδοξία τους. Ε, το σχέδιο που συντονίζει η Λιθουανία με έξι και ε, έξι κράτη-μέλη παρατηρητές που επιτρέψει τα κράτη-μέλη να αλλοβοηθηθούν για να εξασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο ε, ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο και δυνατότητας να αποκριθούν στις προκλήσεις. Ε, βοηθούν επίσης και τις αποστολές ε, ΚΠΑ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ε, Ευρωπαϊκές Ραδιοεπικοινωνίες συντονίζει η Γαλλία για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τα, τους ευρωπαϊκούς στρατιωτικούς ασυρμάτους. Η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας θα μας εξασφαλίσει την διαλειτουργικότητα των στρατιωτικών δυνάμεων στα πλαίσια κοινών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τι εξοπλισμό και τι πλατφόρμες χρησιμοποιούνται και άρα ε, ενισχύεται η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Τα νέα project, ε, ευρωπαϊκή κορβέτα περιπολίας ε, συντονίστρια Ιταλία, θέλει να δημιουργήσει νέα πλοία για να υποστηρίξουν οι τελείως διαφορετικές επιχειρήσεις και αποστολές. Ανάλογα με το είδος των καθηκόντων, ε, που μπορεί να είναι ε, μέτρα κατά της ε, ρήπανσης, ιατρική βοήθεια ή οτιδήποτε άλλο, βοηθούν, βοηθάει αυτή η κορβέτα. Επίσης, έχουμε άλλου τύπου project με τεράστια συμμετοχή 24 από 25 κράτη-μέλη που συμμετέχουν και που δεν θέλουν να δημιουργήσουν ε, δυνατότητες ή τεχνολογίες, αλλά θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν. Ο στόχος είναι να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για να, προχωρήσει, να προωθήσει το συντονισμό για να βελτιώσει τη στρατιωτική κινητικότητα στην Ευρώπη. Στα πλαίσια αυτών των ε, project PESCO θα ήθελα να αναφέρω την στήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα σε αυτά τα project. Ο οργανισμός ε, θέλει να διευκολύνει την ανάπτυξη project για αμυντικές δυνατότητε στα πλαίσια τη μόνιμη διεθνωμένης συνεργασία, ε, Υποστηρίζει όταν τα μελη ε, όταν το ζητήσουν για διάφορα project και τα κράτη-μέλη βασίζονται στην πραγματογνωμοσύνη και την πείρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Προς το παρόν, έξι project PESCO λαμβάνουν ή έχουν λάβει στήριξη ε, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Στήριξη, δηλαδή πραγματογνωμοσύνη αυτό σημαίνει. Και άλλα project τα συζητάει ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα για να τα στηρίξει. Σε ό,τι αφορά το μέλλον, δεν θέλω να πω πολλά, γιατί οι συζητήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί και τα κράτη-μέλη της μόνιμης διαθρωμένης συνεργασίας είναι σε διάλογο. Σε ό,τι αφορά τα project, οι συζητήσεις που γίνονται στα πλαίσια της μόνιμης διαθρωμένης αναθεώρησης θέλει να βελτιώσει τα πράγματα μετά από τη διετή εμπειρία που έχει συσσωρευθεί. Και η γραμματεία της ΠΕΣΚΟ διευκολύνει τις συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχών των κρατών μελών της ΠΕΣΚΟ και θα τα υποστηρίξει για να κάνουν πιθανές αλλαγές στο τρέχον νομικό πλαίσιο τη ΠΕΣΚΟ, δηλαδή τη μόνιμη διαρθωμένη συνεργασία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Σαν Πιέρ Μολνή, τελευταίος. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ο εκπρόσωπος ενός think tank, οπότε ίσως ε, ευχαριστώ κάπως διαφορετικά γιατί τα βλέπω από έξω τα πράγματα και μπορεί να αναφέρθω και σε κάποια ερωτηματικά ε, που γεννούν οι παρεμβάσει των προηγούμενων. Το ΙΡΙΣ είναι ένα δίκτυο εξαμενών σκέψη Think Tank ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο από τη Γαλλία και μας απασχολεί η πολιτική ασφάλειας και άμυνας ε, καθώς και η βιομηχανική αμυντική πολιτική, το δίκτυο ερευνητών και στο πλαίσιο αυτού έχουμε και κάποια έγγραφα τα οποία προετοιμάζουμε για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, ε, του Ταμείου, συγγνώμη, Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ε, και του ΣΠΕΣΚΟ και μιλάμε για τη στρατηγική καθοδήγηση και το πρόγραμμα εργασία που θα πρέπει να εγκριθεί για την περίοδο 2021-2025 μέχρι φέτο το καλοκαίρι. Σε ό,τι αφορά την ε, μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία ΠΕΣΚΟ πρέπει να καταλάβουμε, όπω λέει η Συνδίκη τη Λισαβόνα του 2010, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 2003 και στη Συνθήκη της συνταγματική του 2005. Ε, εκεί υπάρχουν τα σπάργανα. 15 χρόνια όμως χρειάστηκε για να ε, θεσπιστεί αυτή η συνεργασία και όταν αποφασίστηκε να γίνει έγινε πολύ γρήγορα. Είχαμε ένα γερμανογαλλικό διάλογο αρχικά που διευρύνθηκε και όλα αποφασίστηκαν μέσα σε ένα διάστημα τεσσάρων μηνών από το καλοκαίρι του 2017 έως το Δεκέμβριο του 2017. Ένα από τα παράδοξα είναι ότι μάλλον βιαστήκαμε κάπως με την εφαρμογή του μέσου. Έχουμε 20 δεσμεύσει, αλλά ένα από τα θέματα που θα τεθούν πιστεύω όταν γίνει αυτή η στρατηγική επανεξέταση, αναθεώρηση, θα είναι το κατά πόσον αυτά τα commitments, αυτές οι δεσμεύσεις θα μπορούσαν είναι πιο συγκεκριμένες από τις αρχικές 20. Και το δεύτερο, ότι τα 17 project ουσιαστικά είναι αυτά τα οποία είχαν ως στόκ τα κράτη-μέλη. Και κάπως διορθώθηκαν τα πράγματα με τα επόμενα. Σε ό,τι αφορά τις 20 θεσμευτικές αυτές τις υποχρεώσεις. Ε, έχουμε δύο μοντέλα. Συμπληρωματικά κατ' εμέ. Και όχι κατά ανάγκη να ασυμβίβαστα μεταξύ τους. Δημιουργία ευρωπαϊκών δυνατοτήτων είτε εθελοντικά κάποιες χώρες και έχουμε δύο παραδείγματα Φερνίσον Concepts στο ΝΑΤΟ με τη Γερμανία ή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Παρέμβαση της Γαλλίας σε έναν άλλο τομέα και σε διαφορετικό πλαίσιο, όχι ευρωπαϊκό, αλλά είναι θελοντική εδώ η βάση. Οι χώρες που επιθυμούν να κάνουν κάτι μπορούν να το κάνουν. Και όταν δεσμευτούν, το κάνουν χωρίς όμως υποχρέωση. Αυτό είναι το σίγουρο. Και έχουμε την μόνη διαθρομή συνεργασία, ΠΕΣΚΟ, που έχει ένα πλεονέκτημα και ένα ρίσκο. Το πλανήτημα ότι έχουμε αυτές τις δεσμεύσεις που υποχρεώνουν τα κράτη να φέρουν σε πέρα στις δεσμεύσεις τους, αλλά το ερώτημα είναι τι γίνεται εάν δεν το κάνουν. Ένα κράτος δηλαδή, πώς να το πω, θα βγει εκτός πέσκο αν δεν ε, κληρώσει τις δεσμεύσεις του. Θα δούμε τι θα γίνει στα τέλη της χρονιάς. Νομίζω θα πρέπει η διατύπωση να είναι πιο συγκεκριμένη. Σε ό,τι αφορά τώρα την ΠΕΣΚΟ, ε, είναι κάτι που υποτίθεται πρέπει να συμπεριλάνει όλους και καλό θα ήταν να συμβεί αυτό. Θα πρέπει να δεχθούμε πια ότι υπάρχουν και κάποιες χώρες ε, που θα προχωρούν πιο πέρα, στο πλαίσιο μια ΠΕΣΚΟ συν. Αλλά θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί όλοι και αυτό θα, προσπαθ... θα έχει στο κάποιοι να προχωρούν περισσότερο, χωρίς όμως άλλοι να μπουν σε δυσκολίες. Που είναι το θέμα με αυτές τις δεσμεύσεις. Σε ό,τι αφορά αυτά τα έργα, σχέδια, είναι θέμα συνεκτικότητας, συνέπειας, συνολικά σε επιχειρησιακό επίπεδο, επίπεδο δυνατοτήτων. Στις πρώτες δέσμες έργων δεν το είχαμε, το έχουμε στα επόμενα. Αλλά είναι προφανές ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να είναι έτσι πιο εύρωστο το όλο πλαίσιο. Έχουμε τη στρατηγική, έχουμε το επίπεδο φιλοδοξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, πρέπει να το πούμε αυτό, και αυτά πρέπει κάπως να τα συμβιβάσουμε. Δυνατότητες και επιχειρησιακή ικανότητα. Ο Σβέντ Μπίσκοπ, δεν ξέρω, μπορεί να το ξέρετε, είχε συγγράψει ένα πόνημα για τα έργα Πέσκο και έλεγε το κρόκ μήπως θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να δημιουργηθεί ένα project που ουσιαστικά θα περιλαμβάνει και άλλα. σε επίπεδο δυνατοτήτων. Αυτό είναι όμως ε, από κάτω προς τα πάνω, αλλά θα χρειάζεται και να γίνει από πάνω προς τα κάτω. σε ό,τι αφορά το Ταμείο Άμυνας και την ΠΕΣΚΟ. Η ΠΕΣΚΟ είναι πάνω απ' όλα ένα... Είναι κάτι διαφορετικό από το Φορολογικό Ταμείο Άμυνας. Οι στόχοι δεν είναι ίδιοι. Δεν υπάρχει αλληλεπικάλυψη. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο έχει να κάνει με επιχειρήσεις, η ΠΕΣΚΟ σε, απευθύνεται σε κράτη. Δεύτερον, έχουμε τους στόχους του Ταμείου που δεν είναι ίδιοι κατά ανάγκη με αυτή της ΠΕΣΚΟ. Παίρνουν χάρη οι διασυνοριακές συναλλαγές, ε, αποτρεπτικές τεχνολογίες, ε, αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτά είναι βιομηχανικά θέματα. Δεν εντάσσονται στην ΠΕΣΚΟ. Στην ΠΕΣΚΟ, απ' την άλλη, υπάρχουν στόχοι υποσυζήτηση όλα αυτά που λέω βέβαια που είναι πιο πολύ βράχη μεσοπρόθεσμα. Ενώ στο ταμείο υπάρχουν στόχοι που κατ' εμέ είναι πιο μακροπρόθεσμοι. Ιδίως ό,τι αφορά τις τεχνολογίες, τις αποτρεπτικές τεχνολογίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη δυνατοτήτων με ορίζοντα το 2040 και πιο πέρα. Και ένα τελευταίο. Θα πρέπει η ΠΕΣΚΟ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο να διαρθρωθούν, να αλληλεσυνδεθούν. Μία από τις δύο πρωτοβουλίες αφορά την ε, ΚΕΠΑ και η άλλη είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Άρα δεν είναι οι ίδιοι οι κανόνες διακυβέρνησης. Και βέβαια το ερώτημα που πλανάτε είναι η πρόσβαση τρίτων κρατών. Μεταξύ των κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι οι οι απόψει για την σχέση που θα πρέπει να γίνει μεταξύ Πέσκο και Ταμείου Άμυνα. Πολωνία, για παράδειγμα. Μια χώρα σαν την Πολωνία τίνει να αποσυνδέει αυτά τα δύο πιο πολύ. Αν υπάρξει στενή διασύνδεση με το Ταμείο Άμυνας, ε, τίθεται ένα πρόβλημα με το άνοιγμα ε, της Πέσκου σε τρίτα μέρη. Αν όμως πρέπει να χρηματοδοτηθούν έργα απόλυτα συνεπή προς την ιδέα της άνοιξης δυνατοτήτων και ερχόμαστε στο CARD, αυτή τη συντονισμένη αιτήσια πανεξέταση εδώ με τις Σίγουρα κάποιος θα πρέπει να υπάρχει ένα έγγραφο για το, ταμείο, για το επίπεδο φιλοδοξίας ε, που να είναι έτσι μια στέρεη βάση και εκεί θα καθοριστούν όλα αυτά. Απ' την άλλη όμως, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν τα σημαντικότερα έργα και σχέδια. Αυτά όπου η εθνική χρηματοδότηση δεν αρκεί σε ένα συνεργατικό πλαίσιο. Η μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια συνεκτικότητα είναι ότι και τα δύο δημιουργούν συνεργατικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό πραγματικά αλλάζει την κατάσταση, αλλάζει τα δεδομένα. Δεν το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Άρα θέλω να πω ότι ναι, μπορεί κανείς να ασκήσει κριτική και στα δύο και στην ΠΕΣΚΟ που ήδη έχουμε μια διετή εμπειρία. Αλλά τα εργαλεία αυτά και τα δύο είναι καινούρια και απαραίτητα αν θέλουμε να προχωρήσουμε πώς να το πω, σε ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνατότητες στις Ένωσες που είναι πιο αξιόπιστες για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε καταρχάς τον κύριο Σικόφσκι το λόγο. Thank you. <clears throat> I... Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι νέος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε αυτή την επιτροπή, αλλά δεν ε, είμαι νέος στα θέματα τη ΠΕΣΚΟ. Όσον αφορά την τεκμηρίωση όμως είμαι από τους καινούριου. Και ομολογώ ότι δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω όλα όσα ακούστηκαν. Διότι αυτό το οποίο θα ήθελα να γνωρίζω είναι κάτι πολύ απλό. Αν υπάρξει άλλη σύραξη στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα που υπάρχει ένας εθνικιστικός και απρόβλεπτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα είμαστε τόσο προετοίμαστοι όπως ήμασταν στη δεκαετία του 90 στα Βαλκάνια ή θα έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Αν ε, επιδεινωθούν τα πράγματα στη Λιβύη ή στην Αλγερία. Εγώ θα ήθελα να ξέρω τι δυνάμεις και για ποιο διάστημα θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε επιτόπου στο θέατρο των επιχειρήσεων και κατά πόσον μπορούν να επιτευχθούν τα όσα ζητούν οι ψηφοφόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων της ζώνης Σέγγεν από ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να διασχίζουν τα σύνορα. Και θα ήθελα να ξέρω αν η ΠΕΣΚΟ, όπως προτείνεται αυτή τη στιγμή, μας οδηγεί στην εκπλήρωση μιας τέτοιας φιλοδοξίας ή αν θα περάσουμε άλλα, και άλλα χρόνια ή και δεκαετίες κενών συζητήσεων. Θα ήθελα να ξέρω τι ποσά θα χρειαστούν για να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος και κατά πόσον αν οι παρούσες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι προτινόμενες περικοπές αυτές τις προτάσεις αποτελούν απειλή για τα όσα θα θέλατε να επιτύχετε. Νομίζω ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε ευνοϊκά διακείμενοι σε πανευρωπαϊκές λύσεις, τις οποίες δεν μπορούν να προτείνουν τα κράτη-μέλη μεμονωμένα. Και υπάρχει και εμπειρία από τα σφάλματα στην αρχιτεκτονική δομή και τις δυσκολίες στην εξωτερική ανάπτυξη υπό το ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, η χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων από τα κράτη-μέλη και τα ε, αντίθετα ε, κίνητρα τα οποία δημιουργεί για να παραμείνει κανείς εκεί που είναι και να μην αναπτύξει τίποτα. Νομίζω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε μα είχαν πει, ακόμα πριν αναλάβει καθήκοντα ο πρόεδρο ε, Τραμπ, ότι θα υπήρχαν κάποιε επιχειρήσει οι οποίε δεν θα συνέδραμαν. Ε, η Λιβύη βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, γιατί δύο κράτη-μέλη ανέλαβαν να παρέμβουν και θεώρησαν ότι γνώριζαν τι έκαναν. Εμείς φταίμε για το χάλι στο οποίο βρίσκεται και νομίζω ότι θα πρέπει να προτείνουμε και μία ε, αμυντική ένωση η οποία θα αξίζει το όνομά τη. μία αμυντική ένωση που είμαι πεπισμένος ότι θα τύχει ευρεία συνένεση και υποστήριξη από το ευρωπαϊκό κοινό και από πολλά κράτη-μέλη. Αλλά θα ήθελα να τα παρουσιάσουμε όλα με λιγότερο γραφειοκρατικό όρους, με όρους που θα μπορούσα να κατανοήσω εγώ για να μην μιλήσω για τους ψηφοφόρους μου. Θα ήθελα λοιπόν να σας προτρέψω να είστε λίγο πιο τολμηροί, διότι θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Άμυνα είναι μια ιδέα που πλέον έφτασε η στιγμή να ολοκληρωθεί. Έχουμε ηγέτες όπως ο πρόεδρος Μακρόν που προτείνουν να σοβαρευτούμε και αναφέρονται ακόμα και σε ευρωπαϊκό ρόλο, σε πυρηνικούς σχεδιασμούς και πυρηνικές ασκήσεις. Εγώ δεν προτείνω βέβαια η ΠΕΣΚΟ να φτάσει μέχρι σε αυτού του σημείου, αλλά νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχουν βελτιωθεί όσον αφορά την ευρωπαϊκή άμενα και θα ήθελα απλώ να σα πω ότι δεσμεύομαι ότι θα υποστηρίξω τι προτάσει σα υπό την προπόθεση ότι θα είναι πιο τολμηρέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Αρνό Ντανζάν από πλευρά ΣΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, με βάση τα όσα ακούσαμε, δυστυχώς επιβεβαιώνεται η εκτίμησή μου για την Πέσκο. Ναι, μεν όσον αφορά τις αρχές, είναι ένα ουσιαστικό, ενδιαφέρον, σημαντικό βήμα ε, προς τη σωστή κατεύθυνση με πολλές υποσχέσεις όπως ε, το επεσήμανε και ο κύριος Μαλανιές στην ε, αρχική του παρέμβαση αλλά ακόμα πόρο απέχουμε από σημαντικά αποτελέσματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να θεωρήσουμε ότι έχουμε κερδίσει το παιχνίδι αν θέλουμε να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Άμυνα, δεν πρέπει να τα πούμε πολύ γρήγορα και πολύ ε, στεναρά στην κοινή γνώμη, γιατί έχουμε πολλές αρχές, αλλά όχι πάρα πολλά αποτελέσματα από ό,τι άκουσα σήμερα το απόγευμα. Εγώ θα ήθελα να ξέρω σήμερα τι θα γίνει με τα αποτελέσματα, γιατί θα γίνει μια στρατηγική αναθεώρηση ως προς τη διαδικασία. Αλλά τι έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια, πιο συγκεκριμένα τι προχώρησε αυτά τα δύο χρόνια Όλοι θέλησαν να προωθήσουν την ΠΕΣΚΟ. Έχουμε 47, 47 προγράμματα. Ε, κάπου λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και αυτά τα προγράμματα, γιατί δεν είναι και πολύ σοβαρή όλη αυτή η κατάσταση. 47 προγράμματα με πολλές χώρες που προτείνουν προγράμματα, γιατί θέλουν να συμμετέχουν ε, καταρχήν και όχι γιατί περιμένουν και τόσα πολλά συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά τη βελτίωση των ευρωπαϊκών ικανοτήτων. Υπάρχουν λοιπόν και κάποιοι που έχουν και κάποια συγκεκριμένα κίνητρα που εμπνέουν τη συμμετοχή τους. Έχουμε 47 προγράμματα, συμμετέχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πού βρισκόμαστε σε αυτά τα 47 προγράμματα. Πώς επιβιώνουν, πώς προχωρούν. Αυτό που άκουσα σήμερα είναι κάποια ερωτηματικά τα οποία είχαν τεθεί και πριν από δύο χρόνια όταν ξεκίνησε η ΠΕΣΚΟ. Πώ διαρθρώνεται η ΠΕΣΚΟ με την ε, κοινή πολιτική άμυνας. Ναι, θέλω να ξέρω και τι γίνεται και με το ΚΑΡΤ, πώ διαρθρώνεται και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Ναι, πώ διαρθρώνεται η ΠΕΣΚΟ με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Εγώ περιμένω να μου απαντήσετε. Δεν θέλω να με επιβεβαιώσετε ότι θέλετε κι εσεί το ερώτημα. Θέλω να έχω μια απάντηση που θα μπορέσω να δώσω και στου ε, συμπολίτε μου, οι οποίοι τους οποίους τους έχουμε φάει και το κεφάλι δύο χρόνια τώρα και τους λέμε προχωράμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, μην προχωράμε, θα ήθελα να ξέρω κάτι συγκεκριμένο τα κράτη που συμμετέχουν αρχίζουν να ε, έχουν κάποια απτά αποτελέσματα. Εγώ κάτι τέτοιο θα ήθελα να ακούσω και όχι που βρισκόμαστε ως προς τα ερωτηματικά μας, γιατί συμφωνούμε όλοι ως προς αυτά. Όλοι αναρωτιόμαστε πώς θα διαρθρωθεί αυτό το θέμα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Αλλά εγώ περίμενα απαντήσεις και δεν βρήκα απαντήσεις και κάπου απαγοητεύτηκα να συμφωνώ ίσως και με αυτό που είπε και ο Ζανκλέ Μονίκ τελικά ως προς την ουσία. Ναι, έχουμε κάτι θετικό, δεν έχω καμία αμφιβολία περί τούτου, αλλά ο φόβος μου είναι ότι επειδή ακριβώς ε, θέλουμε να έχουμε συμμετοχή όλων και πολύ σημαντικό αριθμό προγραμμάτων και πολύ σημαντικούς ε, ε συμμετέχοντες πέραν των κρατών μελών, Όλα αυτά διαχέονται εδώ και χρόνια σε διαδικασίες και κάνουμε στρατηγικές αναθεωρήσει τη διαδικασία και τελικά από αποτελέσματα ακόμα περιμένουμε και θα περιμένουμε από ό,τι κατάλαβα. Αντιλαμβάνομαι βεβαίω ότι δύο χρόνια δεν είναι μεγάλο διάστημα, αλλά δεν μπορείτε να υποκαταστήσετε εσεί τα κρατημέλη, αυτό το αντιλαμβάνομαι. Θα ήθελα όμω να μου πείτε πού βρισκόμαστε με αυτά τα προγράμματα, τι προχώρησε ποιες χώρες έχουν κάνει ουσιαστικές προόδους, πού έχουμε αυτά αποτελέσματα και πού βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο που έχουμε απλώς ε, ε, σωρία φακέλων πάνω σε ένα γραφείο, αλλά δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Λυπάμαι που είμαι τόσο αρνητικός, αλλά ε, απευθυνόμαστε σε, απευθύνεστε σε ρητούς που πρέπει και εμείς να λογοδοτήσουμε κάπου. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν εχει προχωρησει τιποτα λυπαμαι που ειμαι τοσο αρνητικος αλλα ε σε απευθυνεστε σε ρητους που πρεπει και εμεις να λογοδοτήσω στους ψηφοφόρους μου, στους οποίους είπαμε ότι θα χτίσουμε την Ευρώπη της άμυνας. Ναι, πρέπει τα κράτη-μέλη να κάνουν, το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά υπάρχει και μια γραμματεία ΠΕΣΚΟ η οποία πρέπει να μα πει αν γίνονται κάποια συγκεκριμένα πράγματα ή όχι. Και αν όχι, ε, πέστε μα έχουμε κι εμεί ένα ταπικό ρόλο, ταπεινό ρόλο, μπορούμε ίσω να προωθήσουμε λίγο τα πράγματα. Πρέπει όμω να προσδώσουμε ουσία σε όλα αυτά τα οποία αρχίζουν να συμβαίνουν. Έχουμε ε, δηλώσεις, για παράδειγμα αυτό το Σαββατοκύριακο, από πλευρά του Γάλλου Προέδρου, και τελικά στην ουσία ε, έχουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, από τη μια μέρα στην άλλη μπορούμε να έχουμε και μια τεράστια αποτυχία και εμείς πρέπει να μπορέσουμε να πούμε στους πολίτες μας μην ανησυχείτε ή ανησυχήστε, προχωράει ή δεν προχωράει το πράγμα. Αλλά τώρα εδώ είμαστε μεταξύ μας, στην ευρωπαϊκή μας φούσκα και είμαστε πολύ ε, ικανοποιημένοι για τη στρατηγική αναθεώρηση τη διαδικασία. Ναι, εντάξει να γίνει η στρατηγική αναθεώρηση τη διαδικασία, αλλά δεν βλέπουν επιλύεται το θέμα. Γι' αυτό και απογοητεύομαι. Ευχαριστώ. Πέτρα Οστραβίσιους από το Renew Europe. Ευχαριστώ Ναταλή. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ για να μας ενημερώσατε για την μόνιμη διεθνωμένη συνεργασία, την ΠΕΣΚΟ. Πρέπει να συμφωνήσουμε καταρχάς ότι η συνεργασία αυτή είναι μια σχετικά νέα προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να περιμένουμε θαύματα και μαγεία Αυτό έχει, η συνεργασία αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια, όχι δεκαετίες. Και τα σχέδια τα οποία γίνονται στα πλαίσια της ε, ΠΕΣΚΟ. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του συντονισμού. Γιατί είναι υπόθεση συντονισμού. Και η ομάδα χωρών που συμμετέχουν σε κάποια project PESCO συντονίζονται Παραδείγματο χάρη, το project για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, όπου συντονίζει το project αυτό η Λιθουανία, ο Υπουργό Άμυνα είπε ότι περιμένω την ομάδα που θα φτάσει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη με τα θέματα ε, στον κυβερνοχώρο που αντιμετωπίζουν. Δεν υπήρχε αυτή η ομάδα, τώρα έχει χτιστεί αυτή η ομάδα, υπάρχει μια διαφορετική στρατηγική προσέγγιση και ένα διαφορετικό δυναμικό. Η συμβουλή μου θα ήταν λοιπόν. Θα ήταν μήπω θα έπρεπε να καλέσουμε τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν σε κάποια συγκεκριμένα σχέδια τη ΠΕΣΚΟ και να μιλήσουμε πάνω σε στα συγκεκριμένα project για να καταλάβουμε τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες που διέπουν κάποια project και που είναι πιο προχωρημένα ενδεχομένω από κάποια άλλα. Μπορούμε να καλέσουμε κάποιους ανθρώπους από κάποια κράτη-μέλη και να μπούμε σε λεπτομέρειες για κάθε project. Μπορούμε να μιλήσουμε για ένα ή για δύο, για όσα θέλουμε τέτοια σχέδια, για να καταλάβουμε πραγματικά τις ιδιαιτερότητές τους και τις ιδιαιτερότητες της μόνιμης διαθρωμένης συνεργασίας. Πρέπει να το κάνουμε για να γνωρίσουμε καλύτερα την μόνιμη διαρθωμένη συνεργασία. Όσοι ασχολούνται πάντως με την άμυνα έχουν πολύ θετική άποψη για την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Υπάρχει θετική συνεισφορά από τα κράτη-μέλη και περιμένουν ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο. Τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια θα ακούσουμε πολλά θετικά πράγματα για πολλά σχέδια της ΠΕΣΚΟ. Όταν αυξάνεται ο αριθμός των σχεδίων τα 24 πήγε στα 47, βλέπουμε ότι ε, έχουμε μια πληθώρα σχεδίων, αλλά ελπίζω να υπάρχει και μια εμβάθυνση της συνεργασίας παράλληλα. Με ποιο τρόπο διαχειριζόμαστε την ΠΕΣΚΟ, τη συνεργασία αυτή. Θα αυξήσουμε τον αριθμό των σχεδίων, θα φτάσουμε τα 60 π.χ. Πόσα τέτοια σχέδια πέσκο χρειαζόμαστε, ας πούμε. Μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας. Π.χ. ποιος είναι ο βέλτιστος αριθμός σχεδίων μόνιμης διαρθωμένης συνεργασίας. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλες προτάσεις από τα κράτη-μέλη για να αυξηθεί ο αριθμός των σχεδίων. από τα κράτη-μέλη, τα 27 δηλαδή, και σε ποιου τομεί. Και τα συμπεράσματά σα για το συντονισμό των κρατών μελών, ποια είναι. Βλέπουμε ήδη αποτελέσματα συντονισμού αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν από τις κοινέ διαδικασίες που έχουμε για την λήψη των αποφάσεων, ούτω ώστε η μόνιμη διαρθωμένη συνεργασία να καταστεί ακόμα πιο απρόσκοπτη. Ευχαριστώ ο κύριος Γκάλερ από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τους παρότες, ε, θέλω να τους παρακαλέσω να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο ρωτούμε. Αν είμαστε κάπως επικριτικοί, είναι γιατί θέλουμε αποτελέσματα. Όχι γιατί ε, δεν συμφωνούμε με αυτή την πολιτική, περί το του πρόκειται. Εμεί θέλουμε μεγαλύτερη προστέμενη αξία για την πολιτική και για τα πράγματα τα οποία από κοινού εμείς εδώ θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ε, και υπάρχουν ε, οι αναλύσει ρίσκου και κινδύνου ε, στη Λιβύη, στα Βαλκάνια, στη Βόρεια στο Σαχέλ και οπουδήποτε αλλού. Και από αυτά όλα φαίνεται πόσο αναγκαίο είναι από κοινού να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό να έρθουμε πιο κοντά και νομίζω ότι υπόθηκε και ήταν και ένα σημείο κριτικής ότι πολλά από αυτά τα προγράμματα, τα σχέδια ουσιαστικά βγήκαν από τα σετάρια του εθνικού προγραμματισμού και όταν ε, θεσπίστηκε η ΠΕΣΚΟ ε, κάποιοι σκέφτηκαν ωραία, στα πάμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, μπας και προχωρήσουν ένα ε, αυτό. Επίσης κάτι άλλο που αναφέρθηκε και το θεωρώ και εγώ σημαντικό για παράδειγμα αυτή η διαδικασία κάρτα για την ετήσια επανεξέταση, νομίζω ότι αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει το τι είναι αναγκαίο, τι χρειαζόμαστε, να αναλύσουμε καταρχάς τι έχουμε, πού υπάρχουν ελλείμματα και από εκεί και πέρα, κατά την άποψή μου, νομίζω ότι θα πρέπει με βάση τα συμπεράσματα ε, από αυτή τη διαδικασία να οδηγηθούμε σε ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο πλαίσιο αυτού του CARD για τα διάφορα προγράμματα. Ε, έξι έχουν πάρει το πράσινο φως, αν κατάλαβα καλά. Δεν ξέρω στις λεπτομέρειες τώρα αυτό τι σημαίνει και αν υπάρχει και επαρκή χρηματοδότηση. Ίσως θα μπορούσατε κιόλα ε, να μας πείτε ποια είναι αυτά τα έξι, να μας τα κατονομάσετε. Και κάτι άλλο μια άλλη πτυχή που θέλω να αναφέρω είναι η συμμετοχή των τρίτων κρατών. Υπήρξε μια έτσι κάπως κακή επιστολή από τη ΣΥΠΑ για την συμμετοχή των τρίτων κρατών. Τώρα θα δούμε τι γίνεται και με τη Βρετανία ε, που δεν είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ναι, τότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη συμμετοχή των τρίτων κρατών. Να πρέπει να λύσουμε τα ζητήματα EPR, αλλά να μην υπάρξει εκμετάλλευση. Ε, γιατί εμείς βάζουμε κάποια κονδύλια ε, για κάποιους κοινούς στόχους. Αν παραδείγματο χάρη έχουμε τέσσερα κράτη, ε, τρία από την Ένωση και ένα ας πούμε η Βρετανία, ε, να συμμετέχουν μεν, αλλά να μην παίρνουν ε, από τον υπολογισμό 20-30 δεν ξέρω εγώ πόσο τις εκατό ενώ δεν είναι. Ε, στην Ένωση και θέλουν την ίδια μεταχείριση, δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Θα δούμε και από οικονομικής πλευράς λοιπόν αν αυτό μπορεί να προχωρήσει και πώς ε, θα γίνεται η χρηματοδότηση όταν έχουμε συμμετοχή κάποιου τρίτου κράτους. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπασέσκο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Ας δούμε το αμυντικό μας δυναμικό στην Ευρώπη. Ειλικρινά σας λέω, δεν νομίζω θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα τέτοιο αμυντικό δυναμικό μόνοι μας στην Ευρώπη. Γιατί δεν υπάρχει πυρηνική ισορροπία, Φερρυπίν, με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Παρότι ο πρόεδρος Μακχό είναι έτοιμος να συζητήσει τις πυρηνικές δυνατότητες της Γαλλίας αυτή τη στιγμή. Και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Σαρκοζή, το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας υπέστη μία οπισθοδρόμηση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Ε, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα από το Ντεγκόλ μέχρι να έρθει ο Σαρκοζή όμως. Άλλαξαν τα πράγματα με το Σαρκοζή και την θέση της Γαλλίας στα πυρηνικά. Το θέμα είναι πώς θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μα όταν υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Ας υποθέσουμε ότι τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης πιέζονται από τη Ρωσία. Πώς θα αντιδράσουμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας αυτή τη στιγμή. Η πρότασή μου είναι να εστιάσουμε τις μελλοντικές μας δράσεις σε τρεις άξονες καταρχάς να αναπτύξουμε μια καλή, ένα καλό αμυντικό στρατιωτικό τομέα, μια αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη. Διαφορετικούς εξοπλισμούς και να παράγονται σε διαφορετικές χώρες ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης της κάθε χώρας. Αυτή τη στιγμή όλοι μας παράγουμε, ας πούμε, τάγκς αλλά κάποιο στην Ευρώπη παράγει τα καλύτερα τάγκ. Γιατί θα πρέπει κάθε κράτος μέλο ας πούμε, να φτιάχνει τάγκ. Δεύτερον, δεν θα μπορέσουμε να υπερασπίσουμε την Ήπειρό μα και την Ένωσή μα από τη Ρωσία. Αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα στην Αφρική. Πρέπει να είναι προτεραιότητα αυτό. Γιατί οι απειλές που είναι σχεδόν καθημερινές στην Ευρώπη, είναι από την Αφρική. Παραδείγματο χάρη, στην περιοχή της Αχέλ. Τι γίνεται, μόνο η Γαλλία υπάρχει εκεί. Η Σαχέλ είναι μια τεράστια έκταση και αφήνουμε μόνο τη Γαλλία να τα βγάλει πέρα εκεί πέρα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε Τρομοκράτε που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και μας επηρεάζουν όλους στην Ευρώπη. Ίσως τέτοιε λοιπόν αποστολές θα μπορούσαν να είναι προτεραιότητα για την Ευρώπη. και για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και παρεμβάσεις και για τον Ευρωπαϊκό Στρατό. Δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε την Ευρώπη από όλες τις απειλές. Παραδείγματο χάρη, πρέπει να σταματήσουμε τι επιθετικέ δραστηριότητε τη Ρωσία. Επομένω, θέλω να σα πω, τον αμυντικό κλάδο πώ θα τον αναπτύξουμε. Δεύτερον, σα μίλησα για την Αφρική. Προτεραιότητα και αυτή. Και τρίτον, θα πρέπει να έχουμε ταχύ απόκριση. Είναι σημαντικό αυτό. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια θα ξέρετε όλοι σας φαντάζομαι ότι τα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ και άρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες με εξοπλισμό και στρατό. Αλλά εμείς θα πρέπει να μπορούμε να αντιδρούμε γρήγορα στην Ευρώπη. Αυτή θα μπορούσε να είναι μία αποστολή αποστολές που θα μπορούσαμε να κάνουμε ε, το επόμενο χρονικό διάστημα. Ταπεινή συνεισφορά, αλλά με απτά αποτελέσματα. Ε, σε αυτή τη φάση έχουμε 47 σχέδια. Ε, μπορεί αργότερα να έχουμε 100 σχέδια, αλλά πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Και η προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας από πιθανές απειλές που προέρχονται από την Αφρική. Από το Renew Bernard Guetta. Εντάξει, μ' ακούτε. Τώρα μ' ακούτε. Ευχαριστώ για τη βοήθεια με το μικρόφωνο. Φυσικά και κατανοώ ε, την βιασύνη και την απογοήτευση ενίοτε των συναδέλφων και όχι απλά τη συμμερίζομαι αλλά επαυξάνω γιατί και εγώ βιάζομαι και περιμένω. Αλλά την άλλη πλευρά θυμάμαι πολύ καλά. Πότε ήταν άραγε, πριν από δύο χρόνια περίπου, που και η λέξη Ευρωπαϊκή Άμυνα ήταν σαν προσβολή, σαν βρισιά σε Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα και στο Κοινοβούλιο, αλλά πόσο μάλλον στο ε, Συμβουλίο. Ο κύριο Ντανζά μου κάνει κάτι γκριμάτσε. Τι να πω, τρία χρόνια να πω. Δεν έχει σχέση, δεν έχει σχέση, διότι α κάνουμε τη σύγκριση για να με καταλάβετε καλύτερα. Για να με καταλάβετε καλύτερα. Διότι θα με καταλάβετε καλύτερα, Σα το... Σας διαβεβαιώ. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύγκριση. Πριν λίγο καιρό, στη Βαρσοβία και εκεί ίσω θα συμφωνήσετε μαζί μου και τον Τανζόν, ότι αν λεγόταν, αν κάποιο έβγαζε από το στόμα του τι λέξει Ευρωπαϊκή Άμυνα, ε, θα πάθαιναν αποτροπιασμό κάποιοι. Όχι ο κύριο Σικόρσκι, ο φίλο Μωράντεκ, δεν με εκπλήσει, αλλά και οι πολωνικέ αρχέ σήμερα. Στη Βαρσοβία, την ίδια αυτή πόλη, Ήμουν στο γραφείο του Υπουργού Εξωτερικού πριν από τρει-τέσσερι εβδομάδε και έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή του μιλούσα για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων και με έκοψε και μου είπε: Μα αγαπητέ Μπερνάρ, φυσικά και συμφωνούμε. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Άμυνα. Λοιπόν, όταν υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη, όταν βλέπουμε ότι σήμερα τα μαχητικά αεροπλάνα, τα καλογερμανικό αυτό αεροπλάνο, που κάποιοι το θεωρούσαν αδύνατο. Έχει δρομολογηθεί όταν και τα άρματα μάχησε, αλλά και οι Πολωνοί χτυπάνε στην πόρτα και ανοίγει η πόρτα. Λυπούμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχει αλλάξει η εποχή. Και όταν, αγαπητέ Αρνό Ντανζό, βλέπουμε ακριβώς αυτό που έγινε στο Μόναχο, στη δέσκεψη την ασφάλεια, δεν ήμουν, εσεί ήσασταν από ό,τι κατάλαβα. Α, δεν ήσασταν. με συγχωρείτε. Τέλο πάντων, εγώ δεν ήμουν. Διάβασα όμως τι είπαν οι μεν και οι δε και νομίζω ότι σηματοδοτούν αλλαγή τουλάχιστον στο αφήγημα. Υπάρχει μια γενική ε, αντίληψη, η σφαιρική αντίληψη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις πρωτεύουσε ε, τις ε, πλέον φιλατλαντικές, πώς να τις πω, δεν είναι και ωραία έκφραση αυτή, ας πούμε καταλάβετε τι Ακόμη και σε αυτές τις πρωτεύουσε υπάρχει πλέον η αντίληψη ότι κοιτάνε αλλιώ οι ΙΠΑ τους Ευρωπαίους συμμάχους και αυτό δεν ξεκίνησε επί Τραμπ αλλά και από την πρώτη θητεία Ομπάμα. Και όπως έλεγε η κυρία Μέρκελ στη συνέντευξή της στους Financial Times πριν από κάποιες εβδομάδες είναι δομικές οι αλλαγές αυτές, όχι συγκυριακές. Άρα Μπορεί κανείς να εκφράσει τη λύπη του, να μηδιάσει. Εσείς συνεχώς μηδιάτε, δεν σας βλέπω. Εντάξει, διάστε, αλλά μπορεί κανείς να κάνει κάτι άλλο. Να προσπαθήσει κάτι να προτείνει, να δράσει. Ε, εντάξει, τώρα αυτό δεν χρειαζότανε. Δυστυχώς, σχόλιο εκτός μικροφώνου. Λοιπόν, δεν χρειαζότανε, δεν χρειαζότανε. Αντί λοιπόν να γελάμε ή να θλιβόμεθα, ας σκεφτούμε από κοινού τι μπορούμε να κάνουμε. Συγκεκριμένα, στο Κοινοβούλιο αυτό δεν έχουμε δικαίωμα νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά κανένας δεν μα απαγορεύει να κατεβάσουμε ιδέες και να διατυπώσουμε προτάσεις. Εντάξει, σας πειράζω λιγάκι. Δεν με ακούσατε. Ε, ναι, ακούστε με, ε, αλλά αφού είμαι εδώ τώρα, ακούστε με. Ναι, παρακαλώ, λέει η πρόεδρος, ε, να μην έχουμε γαλλογαλλικό διάλογο. Είναι πολύ συμπαθητικό, μπορείτε να το κάνετε και εκτό, αλλά υπάρχουν και άλλοι που θέλουν το λόγο. Ναι, ωραία. Δύο προτάσει, δύο προτάσεις, λέει ο Γκετά. Νομίζω ότι καλό θα ήταν και άκρο αναγκαίο θα έλεγα, λαμβανομένων υπόψη των γενικών εξελίξεων και τη αλλαγή νοοτροπία στις 27 πρωτεύουσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή η υποεπιτροπή Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και το Κοινοβούλιο συνολικά να σκεφτούν προτάσεις που μπορούν να διατυπώσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μίξερ για το SLD. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι συγκεκριμένος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε μέσω των προγραμμάτων ΠΕΣΚΟ και της ε, Ευρωπαϊκής ε, υπηρεσίε άμυλα και όλα αυτά τα, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυλα και όλε αυτές τι πολύ ωραίες πρωτοβουλίες ε, θα μας βοηθήσει να εξορθολογήσουμε τις διαδικασίες μας, τα πρότυπά μα, να βελτιώσουμε και τη διαλειτουργικότητά μα και είναι όλα πολύ καλά. Όπως το βλέπω εγώ, αρχίζει να αναδύεται ένα μοντέλο όπου ως Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνουμε κάποιους ευγενείς στόχους ε, και κάποιες συγκεκριμένους στρατηγικούς ε, ε, αντικειμενικούς σκοπούς, μια παγκόσμια στρατηγική αν θέλετε, και κάτι αντίστοιχο μεγάλο επίβολο και μετά συνειδητοποιούμε ότι δεν έχουμε και τις δυνατότητες να το κάνουμε. Υπάρχουν σημαντικά κενά στις ικανότητές μας και έχουμε κάποια προγράμματα τα οποία ε, δεν μπορούν τελικά να εκπληρώσουν αυτούς τους μεγαλειώδεις ε, πολιτικούς στόχους. Είναι πολύ σημαντικά και θετικά με όλα αυτά, αλλά όταν ε, φτάνουμε στη χρήση αυτών των ικανοτήτων, διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά μπορεί να αναπτύξει μερικές χιλιάδες εκπαιδευτές και κάποια κράτη-μέλη, λίγα, θα μπορέσουν ουσιαστικά να δώσουν το βασικό όγκο των ε, δυνάμεων με άλλη μορφή. Δεν είναι τεράστιο το πρόβλημα, διότι έχουμε ούτως ή άλλως στην αρχή ε, ενό ελίος συνόλου δυνάμεων και οποιαδήποτε βελτίωση είναι σημαντική, αλλά ως Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συχνά μας περιορίζει η πολιτική ανικανότητα να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Η ερώτησή μου μετά από όλα αυτά είναι ότι συζητήσαμε εδώ πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες ε, για τις ε, ευρωπαϊκές φιλοδοξίες για την επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας. Και αναρωτιέμαι, πιστεύεστε ότι είναι εφικτό αυτό με τις πρωτοβουλίες που έχουμε ήδη αναλάβει ε, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυλας ή πρέπει με επαναστατικό τρόπο να τα βαθμίσουμε όλα αυτά ώστε να επιτύχουμε τελικά αυτή τη στρατηγική αυτονομία. Ευχαριστώ. Η κυρία Λέξμαν από το Έλκη να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μία σύντομη ερώτηση, διότι εξ όσων γνωρίζω και ίσως ε, θα μπορέσω να το επιβεβαιώσει κανείς, αλλά αυτά τα στοιχεία είναι σωστά. Μετά το Brexit, το 80% των δαπανών για την άμυνα εντός του ΝΑΤΟ είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να ξέρω αν αυτό δημιουργεί μια μεγάλη μετατόπιση θα αλλάξει η φύση της συνεργασίας της ΠΕΣΚΟ με άλλα προγράμματα, όπως για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Παρέμβασης, αλλά κυρίως μεταξύ ΠΕΣΚΟ και ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για την ακρίβεια των τελευταίων ερωτήσεων. Να δώσω το λόγο τώρα στους ομιλητές μας για να απαντήσουν ε, για τα θέματα τα οποία τους θέσατε. Εγώ θα ήθελα καταρχάς να πω ότι αυτές οι διαφορετικές ερωτήσεις δείχνουν πόσο ενδιαφέρον υπάρχει για το θέμα αυτό, καταρχάς, και αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει μια διάσταση μεταξύ των πολιτικών φιλοδοξιών και των μέσων που έχουμε στην υπηρεσία αυτών των φιλοδοξιών και μια κάποια απογοήτευση για το επίπεδο ενημέρωσης και πληροφοριών που δίνεται στους ευρωβουλευτές. Σας καλέσαμε εδώ για να μιλήσουμε για την αξιολόγηση, για τα πρώτα βήματα της ε, μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας. Μπορούμε ε, να πούμε από πότε ξεκίνησε η συζήτηση για τα κοινά στρατηγικά μέσα. Έχει ξεκινήσει η συζήτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό ε, και το συζητούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να ξεκινήσουμε κάτι. Τώρα που ξεκινήσαμε, μας λέτε για αξιολόγηση της διαδικασίας και αποφύγατε εσκεμμένα να μην μας μιλήσετε για τη φύση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν τα κράτη-μέλη και κατά πόσον τηρούν αυτές τις δεσμεύσεις ή όχι. Ως προς τα προγράμματα ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δείχνεται κάποιο ενθουσιασμό, τουλάχιστον δεν, ε, δεν έχουμε στην επικοινωνία κάποιο ε, ενθουσιασμό κυρίως ενώπιον των Ευρωβουλευτών που πολύ συχνά εξελέγησαν από ψηφοφόρου που θέλουν να προχωρήσουν τα θέματα της άμυνας. Και όπως και ο κύριος Νταλζάν, όπως και ο κύριος Σικόρσκι, και εγώ πώ θα μιλήσω στου ψηφοφόρους και να τους πω ότι προχωράμε σαφέστατα και με ενθουσιασμό μετά από τη σημερινή συζήτηση. Μου φαίνεται ότι κάνουμε μια από τα ίδια. Ε, μας λέτε ότι, για παράδειγμα, βάζετε μπανάλες σε κυβότια και έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μας για να ξέρουμε ποιο είναι το σωστό ε, μέσο στάθμιση για τι μπανάνε. Συζητάμε θέματα άμυνα σε ένα διεθνέ πλαίσιο στο ε, οποίο έχει αλλάξει με τεράστιε ε, ε, προσδοκίες. Δεν είναι η τελευταία φορά που θα συζητήσουμε βεβαίω τη διαρθρωμένη συνεργασία. Επειδή είναι διακυβερνητικό το θέμα, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το συζητούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι υπάρχουν άμεσε συνέπειε, για παράδειγμα, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο άμυνα και αυτό αφορά φυσικά τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε κάποια πράγματα περισσότερο, να είστε πιο σαφεί μαζί μα, διότι περιμένουμε να ξέρουμε κάποια πράγματα και αν δεν λειτουργεί κάτι, πρέπει να στραφούμε προ τα κράτη-μέλη που δεν κάνουν απαραίτητο αυτά που λένε ε, στις ε, ε, δηλώσεις τους. Δεν ξέρω ποιο θέλει να πάρει πρώτο το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλες αυτές τις παρατηρήσεις, ο κύριος Μολενάρ. Βεβαίω είμαστε εδώ για να σα δώσουμε ό,τι πληροφορία θέλετε και να απαντήσουμε σε όποια ερώτηση έχετε. Και λυπάμαι αν ήταν σε πολύ τεχνικό επίπεδο τα όσα είπα και δεν ήταν επαρκώ πολιτικά. Εμεί είμαστε αυτοί οι οποίοι ασχολούμαστε με τι λεπτομέρειε και ε, απαντούμε όλε αυτέ τι διεξοδικέ ερωτήσει που προσπαθήσαμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα. Φυσικά είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό η στρατηγική αναθεώρηση τη ΠΕΣΚΟ και προσπάθησα να αναφερθώ στη στρατηγική, πολιτική και οικονομική αξία τη δουλειά που πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Ταυτόχρονα όμω, είμαστε και στα σπάργανα τη διαδικασία. Τώρα αρχίζουν αυτέ οι συζητήσει. Δεν έχουμε λοιπόν όλε τι απαντήσει ακόμα, αλλά μπορώ να σα πω ότι η ΠΕΣΚΟ μαζί με το Ταμείο Άμυνα και με την ΚΑΡΤ αποτελούν μέχρι τώρα την καλύτερη απάντηση για τη δημιουργία πραγματικά μιας Ευρωπαϊκής Άμυνας. Όσον αφορά τα διορθωτικά ζητήματα που ε, αντιμετωπίσουμε, το 80% της δαπάνης για την άμυνα είναι σε εθνικό επίπεδο ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι πολλαπλασιάζονται τα αμυντικά συστήματα και η βιομηχανία και αυτό σημαίνει ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, ακόμα δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τα καθήκοντα τα οποία έχουμε θέσει για 20 χρόνια. 60.000 στρατεύματα σε 60 μέρε. Αυτό είχαμε προβλέψει όσον αφορά την ε, παρέμβαση στα Βαλκάνια ε, τότε στη δεκαετία του 90. Ακόμα δεν μπορούμε να απαντήσουμε αποτελεσματικά και να έχουμε τέτοια ανάπτυξη. Προσπαθούμε βεβαίως να τελειοποιήσουμε και να αξιολογήσουμε τους στόχου αυτούς, αλλά ε, μία επιφύλαξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει ε, επιλεκτική άμυνα ή εδαφική άμυνα, αυτή είναι η εδαφικη αμυνα αυτη ειναι δουλεια του ΝΑΤΟ. Οι ικανότητε που αναπτύσσουμε που ε, αναπτύσσουν τα κράτη-μέλη και διαθέτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τι επαφέ του. Αυτά που κάνουμε λοιπόν μπορεί να βοηθήσουν και τον ΝΑΤΟ. Όσον αφορά τι προτεραιότητε, είναι ε, σημαντικό το ζήτημα γιατί συλλογικά δεν έχουμε τα χρήματα ω ε, κράτη-μέλη ή ω Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα να χρηματοδοτήσουμε τα πάντα. Επομένω πρέπει να ιεραρχήσουμε τι προτεραιότητε για να ξέρουμε βέβαια ποιε θα είναι οι προτεραιότητε. Δεν μπορώ εγώ να το προβλέψω, αλλά σίγουρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε να μπορούμε να διεξάγουμε τις επιχειρήσεις που θα πρέπει να διεξαχθούν όταν έρθει η ώρα, είτε είναι στην περιφέρεια της Ευρώπης, είτε στην Αφρική, να μπορέσουμε λοιπόν να <clears throat> παρεύουμε πράγματι όπως και παράδειγμα στη Λιβύα. Έχουμε δυνάμεις στην Ευρώπη, αρκετές θα μπορούσα να σας απαντήσω, αλλά το θέμα είναι τα θέματα επιμελητίας, ε, τις ικανότητες, όλα αυτά πώς μπορούμε να τα έχουμε και να έχουμε συνεργασία σε δύσκολο και επικίνδυνο περιβάλλον. Θα απαντήσουν βέβαια και οι στρατιωτικοί συνάδελφοι από αυτού. Υπάρχει ένα σύστημα για να εξετάσουμε όλε αυτέ τι εκδοχέ και να δούμε πού θα πρέπει να επικεντρωθούμε, αλλά είναι χρονοβόρο και δεν είναι κάτι το οποίο είναι στα δικά μου τα χέρια θα ήθελα και εγώ να διαβιβάσω το πάθος σας στις συζητήσεις που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και πιστεύω και εγώ ότι η ώρα, το στρατηγικό πλαίσιο είναι σαφές, υπάρχει στρατηγικός αντίκτυπος στην Ευρώπη, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θα είναι μαζί μας σε κάθε βήμα, επομένω πρέπει να είμαστε πιο αυτόνομοι. Η στρατηγική αυτονομία ως όρος χρησιμοποιείται λίγο αφιδώς, ε, είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να βελτιώσουμε βεβαίως και προσπαθούμε να το κάνουμε σε ανταλλαγή μυστικών πληροφοριών, ανάπτυξη ικανοτήτων και ούτω καθεξής. Τη σήμερον ημέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφορά μόνο τις δυνάμεις που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά προστασία, εξωτερική, εσωτερική διάσταση, ε, διεθνείς απειλές ε, και φυσικά πρέπει να κερδίσουμε, λέει κάποιος από τη λομή γίνεται ναι, φυσικά πρέπει να κερδίσουμε και πρέπει να είμαστε μπροστά στο παιχνίδι, να μην μείνουμε πίσω. Συμφωνώ λοιπόν ε, και πρέπει να σας χρησιμοποιήσουμε ως πηγή έμπνευσης και ζητώ συγγνώμη. Τώρα, αν ήταν κενά τα όσα κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια, νομίζω όχι. Για πρώτη φορά έχουμε νέα εργαλεία, τα οποία δεν θα μπορούσε να διανοηθεί κάποιο καν πριν από τρία-τέσσερα χρόνια. Και φυσικά υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα για το, στον προπολογισμό για την άμυνα. Υπάρχει Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. Ε, βέβαια, προσβλέπουμε σε φιλόδοξη ε, χρηματοδότηση και μα ανησυχούν αυτέ οι περικοπέ που είδαμε, αλλά για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υπάρχουν οικονομικά κίνητρα για να σταματήσει αυτό το αδιέξοδο στο οποίο είχαμε περιέλθει τόσα χρόνια και ώστε η ευρωπαϊκή ε, συνεργασία στην άμυνα να μπορέσει να προχωρήσει. Το κατά πόσο θα προχωρήσουν τα πράγματα καλύτερα αν έχουμε ένα ε, επιχειρησιακό σενάριο εξωτερικής παρέμβασης, δεν ξέρω, θα πάρει 5 έως 10 χρόνια και φυσικά αυτό είναι αυτό το οποίο θα ε, πω εγώ στη συζητήση με τα κράτη-μέλη και οι συνάδελφοι μαζί μου να επικεντρωθούμε σε τέτοια αποτελέσματα και να δούμε ότι σταδιακά σε 5-10 χρόνια από τώρα θα είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τι επιχειρήσει που θέλουμε. Όσον αφορά του φορολογούμενου, νομίζω ότι το σημαντικό μήνυμα είναι να ε, δώσουν χρήματα τα οποία θα του αποφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξία. Να μην διαχέονται τα χρήματά μα, να τα κάνουμε από κοινού και να επικεντρωθούμε στα όσα χρειάζεται η Ευρώπη και τι μπορεί να παρέχει η βιομηχανία και όχι ότι θέλει να παρέχει. Ε, θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση λοιπόν η οποία θα πρέπει να ε, παρακινείται από τις ικανότητές μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είχαμε προτεραιότητες για την ανάπτυξη ικανοτήτων οι οποίες αποτελούν και το κινητήριο μοχλό για όλες τις διάφορες πρωτοβουλίες. Επικεντρωνόμαστε σε ίδιους τομείς. Οι στρατογικές ελλείψεις συμπεριλαμβάνονται εδώ για να επικεντρωθούμε και στους κατάλληλους τομεί. Έχουμε μια σειρά από πιο τεχνικά, αν θέλετε, ε, στοιχεία για να απαντήσουμε στο πώς ε, έχουμε τη διάδραση των διαδικασιών, έχουμε τις διάφορες επιτροπές και παρακολουθούμε και τα χρονοδιαγράμματα. Και ζητώ συγγνώμη αν φάνηκε ότι απλώς τώρα τα ανακαλύπτουμε σιγά σιγά. Είναι αυτά που κάνουμε κάθε μέρα. Αυτό που μπορούμε σίγουρα να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τα πράγματα και να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα που θέλουμε στη συνέχεια. Η ΠΕΣΚΟ είναι και νέα ως προς αυτή την έννοια, διότι τελικά τα κράτη-μέλη θα πρέπει το καθένα να αποδείξουν ότι τηρούν τις δεσμεύσεις τους και μετά μέσω της αξιολόγησης γραμματείας της ΠΕΣΚΟ, εάν δεν τις τι στηρούν τι δεσμεύσει του, μπορούμε να το δείξουμε και να υπάρχουν κάποιε κυρώσει βάσει τη συνθήκη που θα επιτρέψουν, για παράδειγμα, αναστολή τη ε, ιδιότητα του μέλου. Δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο στην πράξη, αλλά για πρώτη φορά υπάρχει και αυτή η δυνατότητα στο πλωστάσιό μα που δεν είχαμε στο παρελθόν. Αν μπορούσα να κάνω και μια προσωπική παρατήρηση, εγώ ήμουν πρόεδρο ομάδα εργασία στο Συμβούλιο τη πολιτική και στρατιωτική ομάδα που ανέπτυξαν όλα αυτά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Οι συζητήσει που κάναμε το 2013 σε σχέση με το πού βρισκόμαστε τώρα ε, είναι χιλιόμετρα μπροστά. Το θέμα της άμυνας ήταν θέμα. Η συνεργασία για την άμυνα ήταν σημαντικό πρόβλημα. Τώρα συζητούμε για συνεργασία στην άμυνα. Έχουμε προχωρήσει πολύ λοιπόν. Βέβαια, το κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετική προσέγγιση και διαφορετική προοπτική αυτό το είπε και ο υπατό εκπρόσωπο Μπορέλ όταν εξετάζουμε την Ευρώπη. Φυσικά όλα τα κράτη-μέλη δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα και ενδιαφέροντα για την ασφάλεια, την ίδια ιστορία και την ίδια προσέγγιση. Και εδώ αυτή η λεγόμενη στρατηγική πηξίδα θα είναι πολύ σημαντική, γιατί θα είναι ένα έγγραφο το οποίο θα βασίζεται σε στρατηγικό επίπεδο και σε μια ανάλυση η οποία θα γίνει συλλογικά, ώστε να έχουμε μια κοινή εικόνα για τις απειλέ και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια κοινή στρατηγική νοοτροπία στη συνέχεια. Και εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω και με κάποιους από τους ευρωβουλευτές, πρέπει να μειώσουμε το κενό μεταξύ φιλοδοξίας και δράσης και αποτελεσμάτων. Να, όχι να μειώσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας απαραίτητο, αλλά να είναι πιο σταδιακό και πιο ρεαλιστικό στην προσέγγιση μας και στον τρόπο με τον οποίο επιτυχάνουμε τα όσα έχουμε καθορίσει ότι θα κάνουμε. Πολύ ευχαρίστω να συνεχίσω βεβαίω και τη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή σα, κυρία Πρόεδρε, και να απαντήσω σε όποια ερώτηση έχετε επί του θέματο. Η ΠΕΣΚΟ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο και δίνει συγκεκριμένε πολιτικέ δεσμεύσει και υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν εκθέσει. Ε, δεν συνέβαινε αυτό στο παρελθόν. Ε, Εμεί ελέγχουμε τι εκθέσει. Τώρα πρέπει να γίνει καλύτερη διαχείριση για να δούμε πού μπορούμε να έχουμε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους στόχους που θέτουμε. και φυσικά να προχωρήσουμε προς τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πολύ σωστά λύσατε. Αυτά νομίζω. Πολύ ευχαρίστως βέβαια να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Um... Ευχαριστώ. Οι υπόλοιποι πολύ σύντομα δύο-τρία λεπτά έκαστο. Γιατί έχουμε και ένα άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη αμέσω μετά και έχουμε λιγάκι καθυστερήσει. Βλέπετε πόσο ενδιαφέρον όμω έχει για μα αυτό το θέμα. Και μα ενδιαφέρει βεβαίω το να ακούσουμε πράγματα από εσά. Έτσι αυξάνεται και το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Σωστές ερωτήσεις, θα έλεγα. σε σχέση με αυτά που ρωτήσατε για το αν μπορούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τα Δυτικά Βαλκάνια. Έχει ήδη απαντηθεί εν μέρη το θέμα αυτό. Αλλά η απάντηση είναι σαφής. Δεν έχουμε τις δυνατότητε που θα μας επιτρέψουν στα σοβαρά να κάνουμε τέτοιου επιχειρήσει στα Δυτικά Βαλκάνια. Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, ξέρουμε ακριβώ τι μα λείπει. Έχουμε διάφορα σενάρια σχεδιασμού που συμπεριλαμβάνουν και τα Δυτικά Βαλκάνια και τώρα προσπαθούμε να καλύψουμε αυτά τα κενά σε ό,τι αφορά τις δυνατότητές μας. Έτσι δρομολογείται μια συνεργασία ΠΕΣΚΟ. Από εκεί ξεκινάμε το σχεδιασμό. Και τα ελλείμματα οφείλονται σε δύο πράγματα. Αν ζητήσετε από τα κράτη-μέλη, έτσι, από τη μία στιγμή στην άλλη, να ετοιμάσουν ή να παρουσιάσουν κάποια project, ε, εξετάζουν τα εθνικά του σχέδια, τα οποία γίνονται για 5, 10 ή 15 χρόνια. Δεν μπορείτε να περιμένετε μεγάλα κενά ε, στα εθνικά σχέδια τα οποία θα μπορούσαν να καλυφθούν με project PESCO. Επομένως θα πρέπει να έχουμε το βλέμμα στραμμένο πιο πολύ προς το μέλλον. Τώρα αρχίζει να κινείται το πράγμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Όντως ε, εξετάζουμε, έχουμε το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, στηρίζουμε τα κρατημέλη, στηρίζοντας τα κατάλληλα σχέδια, τα κατάλληλα προγράμματα, τώρα συνειδητοποιούμε ότι η τελευταία παρτίδα σχεδίων ήταν πολύ πιο εύκολο να υλοποιηθούν και εστιάζονταν στις ανάγκες παρά η πρώτη παρτίδα, ας πούμε. Επομένως, προχωράμε. Ο δεύτερος λόγος ελλείψεων, και αυτή είναι η προσωπική εκτίμηση, είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε τι σκοπό έχει αυτή η μόνιμη συνεργασία. Γιατί γίνεται. Γίνεται κυρίως για να διατηρήσουμε τον ευρωπαϊκό στρατηγικό, την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία ή κυριαρχία ή θέλουμε να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη στο να αναπτύξουν περαιτέρω τις ε, δυνατότητές τους. Μερικά κράτη-μέλη έχουν το βλέμμα στραμμένο στο ΝΑΤΟ, και άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι κάνουμε ακριβώς με την ΠΕΣΚΟ. Οι προτεραιότητες μας είναι ευρύτερε από την ΚΠΑ. Ξεπερνάμε τα πλαίσια της ΚΠΑ. Και αυτό σημαίνει ότι τα κενά δυνατοτήτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, αμυντικών δυνατοτήτων ή στατιωτικών δυνατοτήτων, λαμβάνονται υπόψη, αλλά δεν είναι, δεν κολλάμε σε αυτά απλώς. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί. Δηλαδή, τι κάνει η ΠΕΣΚΟ τελικά. Τι σκοπό έχει, γιατί υπάρχει. Και κλείνοντα θα ήθελα να μιλήσω για ένα project της ΠΕΣΚΟ, που θα ήθελα να το κοιτάξετε πιο προσεκτικά. Για, το, για τις επιχειρήσεις ε, ανταπόκρισης σε κρίσεις. Αυτό είναι ένα project που θα μπορούσε βραχυπρόθεσμα, ε, μακροπρόθεσμα, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή δύναμη η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας. Αυτή τη στιγμή το συζητάμε με τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη για να προχωρήσει, να δρομολογηθεί αυτό το project. Βασικά αυτά κάνουμε. Ευχαριστώ. Και οι δύο τελευταίοι ομιλητέ. Ο καθενα ετσι έτσι δύο-τρία λόγια να πει για να κλείσουμε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος και να απαντήσω παράλληλα όσο μπορώ. Εμείς ε, κοιτάμε και τις λεπτομέρειες βεβαίως, αλλά η ΠΕΣΚΟ δεν είναι το μαγικό ραβδάκι είναι παρόλα αυτά ένα πολύ δυνατό εργαλείο που έχουν τα κράτη-μέλη. Αν δούμε το προσδόκιμο ζωής ενός ανθρώπου, τι είναι, 82-83 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω. Ας δούμε όμως την ε, Πέσκο που είναι μόνιμη και ας ξαναδούμε μετά από δύο χρόνια τον, τον άνθρωπο. Μετά από δύο χρόνια ένας άνθρωπος ε, θα, για να αν συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό θα μπορέσει να τον κερδίσει, πρέπει να είναι προετοιμασμένο. Επίση, δεν μιλάμε μόνο για έναν άνθρωπο που. ένα δρομέα, α πούμε. Εδώ είμαστε. Μιλάμε για μια ομάδα ράγκμπι. Μέσα σε δύο χρόνια δηλαδή, τα κράτη-μέλη δημιουργούν συνεργασία και παίζουν αγώνες ράγκμπι γιατί έχουν ομάδα, άρα συνεργάζονται. Άρα υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία ήδη στο ενεργητικό τη ε, ΠΕΣΚΟ. Γιατί με ρωτήσατε τι επιτυχίε έχει. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία καταρχά. Αν δούμε τα, τα project ε, ΠΕΣΚΟ, το είδο τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, αυτό το είδο της συνεργασια τελειως τελείως νέο. Υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν ήταν ε, συνηθισμένα να συνεργάζονται με άλλε ομάδε κρατών μελών και τώρα συμμετέχουν σε τέτοια project ΠΕΣΚΟ. Κοιτάξτε την ιστοσελίδα πολύ προσεκτικά που είναι προσπελάσιμη στο κοινό pesco.europa.eu ε, και κοιτάξτε τι συνεργασία έχουν τα κράτη-μέλη. Ένα σχέδιο, ένα project μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Τα κράτη-μέλη δεν, μπορούν, δεν χρειάζονται την ΠΕΣΚΟ για να προχωρήσουν ένα σχέδιο, να το υλοποιήσουν. Αλλά η ΠΕΣΚΟ επιτυχάνει κάτι άλλο. Κάνουμε μαζί σχεδιασμό καταρχάς. Οι στρατιωτικοί αρχίζουν να συνεργάζονται από το ένα κράτος μέλος με τους στρατιωτικούς του άλλου. Ε, πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό ένα στρατιωτικό, ένα στρατιωτικό πλαίσιο και ένα χρονικό ορίζοντα για να υπάρχει, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια σύγκληση. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για να επικοινωνήσουν καλύτερα. Γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη, Γιατί η ΠΕΣΚΟ είναι δημιουργία των κρατών μελών. Έχουμε μία ε, γραμματεία που την αλλά τη θέληση για να κάνουν τέτοια πράγματα μαζί την έχουν τα κράτη-μέλη. Τώρα για το ερώτημα για το ΝΑΤΟ. Ε, στα πλαίσια της κοινή δήλωση. Ε, θέλουμε να κάνουμε κοινέ προσπάθειες και να έχουμε και κοινά αποτελέσματα. Βοηθάμε τα κράτη-μέλη να φτάσουν σε κοινά αποτελέσματα με βάση αυτήν την κοινή δήλωση. Και μετά από αυτά τέλειωσα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μολνή τρεις φράσεις σας δίνω. Πολύ σύντομα. Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσει των Ευρωβουλευτών σε ό,τι αφορά τις φιλοδοξίες. Πάρα πολύ θετικά, ναι, αυτά. Δεύτερον, να σας πω ότι ακόμα και εγώ διερωτήθηκα. Μήπως εγώ πλήττομαι από τον ιό της, του ευρωσκεπτικισμού ή ε, της σκληρής και ξύλινης γλώσσας, ας πούμε, της γραφειοκρατίας. Όχι, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Στην ΠΕΣΚΟ, οι 20 δεσμευτικές οι 20 δεσμευτικοί στόχοι. Πρέπει να τους γράψουμε εκ νέου. Γιατί κάποια στιγμή υποχρεώσεις υπήρχαν, 20% ε, επενδύσεις, δαπάνες επενδύσεων και τα υπόλοιπα ήταν εγώ θέλω να είμαι νέος όμορφος και υγιής. Κανένας δεν μπορεί να πει τίποτα αντίον αυτού. Το θέμα είναι στο εθνικό σχέδιο εφαρμογής αν τα κράτη-μέλη σέβονται τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες δεν είναι και πολλές, είναι αρκετά ήπιες, για τα 47 project. Ποιο είναι το πρόβλημα, από τι πάσχουμε. Έχουμε ένα επίπεδο φιλοδοξίας έτσι λίγο αόριστο στη διατύπωση και από πίσω δεν υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός με ομάδες ε, στρατηγικών λειτουργιών, ας πούμε, όπως κάνουμε στη Γαλλία. Απλώς προσπαθούμε να ε, έχουμε προσέγγιση των στρατηγικών εγγράφων. Αν είχαμε πέντε, ας πούμε, στρατηγικές ε, λειτουργίες ή στόχους, θα ήταν πολύ πιο σαφή τα πράγματα και θα προχωρούσαμε με τα project που ήταν σημαντικά, θα καταργούσαμε αυτά που δεν προχωρούν ε, και θα είχαμε πολύ λιγότερα από 47 project. Για τους Γερμανούς έχουν δύο project που είναι ακριβώς τα ίδια. Ε, ε δικά τους εθνικά project που είναι ίδια ακριβώ με τη ΠΕΣΚΟ. Το θέμα είναι πώ θα μπορέσουμε να κάνουμε μια σύγκληση αυτών των κοινών σχεδίων. Γιατί υπάρχουν επικαλύψει περιτέ. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να καταργηθούν. Εάν παρουσιάσουμε αυτά τα πράγματα πολύ πιο σαφώ, λέγοντα να τα αποτελέσματα, να τι θα δώσουμε, να τι θα προκύψει, όλα θα είναι πιο ξεκάθαρα και για το μυαλό των Ευρωβουλευτών, αλλά και στο μυαλό των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Πολύ ενδιαφέρον ε, είδατε ότι υπάρχει. Μεγάλη στήριξη. Περιμένουμε όλο και πιο ενδελεχεί συζητήσεις, όχι γιατί δεν μας αρέσει η ΠΕΣΚΟ, απλώς γιατί θέλουμε να επιτύχει. Επομένως, για να κλείσουμε αυτό το τμήμα των συζητήσεων μας, θέλω να σας πω απλώς ή στο επανειδήν. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημίσιας διάταξης, το Brexit αυτό το σημείο θα το συζητήσουμε και κλεισμένο των θυρών. Και οποιοδήποτε δεν ε, έχει εξουσιοδότηση να συμμετάχει σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να αποχωρήσει από την αίθουσα. Θα ξαναρχίσουμε σε δύο λεπτά και συγγνώμη για την καθυστέρηση.